και της καταπολέμησης των μη μεταδοτικών ασθενειών παγκοσμίως. Σας ευχαριστώ για την πολύ αποδοτική συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε, Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Πράγματι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και από στατιστική πλευρά και από κοινωνιολογική πλευρά πρέπει να σημειώσουμε ότι από τι 18 παρεμβάσει οι 13 προέρχονταν από γυναίκε συναδέλφου. Και φυσικά όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα τέτοιου ε, χαρακτήρα, τέτοια σημασία, φαίνεται ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένε και δεσμευμένε οι γυναίκε από του συναδέλφου άντρε στο θέμα αυτό. Και θέλω να τη συγχαρώ γι' αυτό. Έχω λάβει δύο προτάσει ψηφίσματο ε, που θα κλείσουν και αυτή τη συζήτηση. Η ψηφοφορία από αυτόν θα λάβει χώρα σε λίγο από τι 12 και μετά. Επόμενο σημείο στην ομιλητική διάταξη. Προσφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πολιτική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη τη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών που θα πραγματοποιηθεί το 2012. Διάσκεψη τη ITU. Είναι μια προφορική ερώτηση από την Επιτροπή Βιομηχανία Έρευνα και ενέργεια. Ο συνάδελφο Ρόιλ έχει το λόγο, ο οποίος και θα υποβάλει ως συντάκτης ε, την προφορική ερώτηση. Έχετε πέντε λεπτά για την παρέμβασή σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία ε, ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το, τη διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών της CTU του 2012 που αναγνωρίζει και τονίζει ότι τα κράτη-μέλη είναι ανεξάρτητα μέλη της CTU αλλά πολλά θέματα έχουν ευρωπαϊκή σημασία και εδώ θα αναφερθώ σε ορισμένα τα οποία άλλωστε αναγνωρίζονται και στην ημερήσια διάταξη δηλαδή την διασυνοριακή ε, ε, ε, επιρροή των ψηφιακών επιδόσεων, των, της διαστημικής πλοήγησης που είναι σημαντικό για το Γαλιλαίο ή το θέμα της εισαγωγής ε, ε, συγχρόνων συστημάτων ε, που έχουν σημασία για την διαχείριση των αεροπορικών συγκοινωνιών ή τα διάφορα αμ ε, ε, θέματα των μικρών ε, κινητών συσκευών που έχουν σημασία για την ιατρική και για άλλους τομείς. Άρα τα θέματα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν έχουν άμεση επιρροή σε πολλούς τομείς της εσωτερικής αγοράς αλλά και τη διεθνή πολιτική και την πολιτική του διαστήματος και ως εκ τούτου πρέπει να επέμβουμε εις ε, τις ε, διεθνείς επικοινωνίες ε, και δίδεται στη διάσκεψη αυτή μία νέα διάσταση που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής. Η Επιτροπή μας λοιπόν αναρωτήθηκε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίσει τις ευρωπαϊκές ιδιομορφίες εις την διάσκεψη αυτή και να δηλώσει ότι η Ευρώπη μιλάει με μία φωνή στα σημαντικά αυτά θέματα διότι υπάρχουν πολυμερείς συζητήσεις όπου παρουσιάζονται διάφορες απόψεις και ε, τουλάχιστον η χρήση των συχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιαστεί σωστά στην ETU αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό και διατυπώσαμε τη θέση αυτή διότι επιπλέον στο συνέδριο αυτό πρόκειται να καθοριστούν συζητηθούν τα θέματα για την επόμενη διάσκεψη όπου θα εξεταστεί ο αναβαθμισμένος χαρακτήρας Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα πλαίσια της παγκόσμιας αυτής διάσκεψης ως εκ τούτου ε, θεωρήσαμε ότι υπάρχουν θέματα που είναι σημαντικά και ένα από τα πιο σημαντικά είναι κάτι το οποίο έχει σημασία με, ε, την, ε, με την θέση στο φάσμα των 800 MHz και γι' αυτό σας υπενθυμίζω την έκθεση του κυρίου Χακμαρτ πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσμακος. Ήταν μια έκθεση η οποία έγινε αποδεκτή με μεγάλη πλειοψηφία όπου ε, εξετάζαμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τα ψηφιακά δεδομένα σε μια συχνότητα η οποία μπορεί να προωθήσει τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί ε, να επιτύχει τις ε, κινητές ε, μεταδόσεις στοιχείων. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ καινοτόμα θέματα αλλά να εξασφαλίσουμε ότι όποιος χρησιμοποιεί αυτές τις συχνότητες αυτές να αναγνωρίζει τι ρόλο διαδραματίζει και στην περίοδο κρίσεως συνήθως λέμε τι δεν πάει καλά και που έχουμε προβλήματα. Πρέπει λοιπόν όταν έχουμε προωθήσει ένα θέμα και είναι παραγωγικό να μπορούμε μπορούμε να το διακηρύξουμε και στη διάσκεψη αυτή μας δίνεται αυτή η ευκαιρία και γι' αυτό υπάρχει η επερώτηση ε, για να μπορέσουμε να τονίσουμε ε, στην παγκόσμια αυτή διάσκεψη περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Χέκμαρκ θα αναφερθεί και περαιτέρω στο θέμα αυτό για τις δυνατότητες των συχνοτήτων που μπορεί να επιτρέψει η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη διότι δεν έχει έχει λόγο να μιλάμε για ανάπτυξη και όταν μας δίδονται οι ευκαιρίες να μην τις εκμεταλλευόμαστε. Εξού και το προφορικό ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ την Επιτροπή Ήτρε διότι έθιξε αυτό το ζήτημα και το έθεσε στην ημερήσια διάταξη. Τα πιο σημαντικά ζητήματα αφορούν τον συντονισμό του ψηφιακού μερίσματος στα 800 MHz και επίσης το ραδιόφασμα όπως θα οριστεί στην εσωτερική αγορά. Εδώ ήδη υπάρχει νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν λάβουμε υπόψη την ολοένα και μεγαλύτερη συνένεση και με βάση την παγκόσμια διάσκεψη ραδιο, επικοινωνιών, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να, ε, να προωθήσουμε περαιτέρω διευθετήσεις σε αυτή την ανακοίνωση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν πλήρως έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα το οποίο θα άλλαζε τα, τους εσωτερικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να υποπτεύσουμε αυτό το πλαίσιο και αν τα κράτη-μέλη δεν συμμορφωθούν τότε η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης θα προωθηθούμε, θα επεκταθούμε, με συγχωρείτε, πέρα από αυτή την ad hoc προσέγγιση και θα επανεξετάσουμε και το ενδεχόμενο τέλος του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ITU. Με βάση την διάσκεψη του 2015 θα δούμε πώς θα κινηθούμε με βάση την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών 2012 με βάση την, ε, ε, ε, την ευρυσυχνότητα. ευρυζωνικότητα, με συγχωρείτε. Και αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε έναν απογραφικό κατάλογο ραδιοφασμάτων, κάτι το οποίο αφορά το γενικότερο πρόγραμμα ε, ραδιοφάσματος, το οποίο εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να ε, φτάσουμε σε περαιτέρω βήματα σε σχέση με την τυποποίηση αυτού του προγράμματος. Τώρα θα λάβουν το λόγο εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων οι ομιλητές, ο κύριος Χέκμαρκ για δύο λεπτά εξ του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την απάντηση που έδωσε στην προφορική ερώτηση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά όταν συζητούμε το θέμα αυτό. Φάσμα πρώτον. Όταν μιλάμε για φάσμα μιλάμε για τηλεπικοινωνίε. Ε, για κινητό ασύρματο δίκτυο, διάφορε συσκευέ, τεχνολογίε. και νομίζω ότι είναι ένας από τους τομείς ε, στην παγκόσμια κοινότητα που αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς. Λέω παγκόσμια κοινότητα γιατί δεν μιλάμε μόνο για την οικονομία, μιλάμε για την πολιτική, μιλάμε για τις πληροφορίες, την επιστήμη και πολλούς άλλους τομείς της κοινωνίας. Πράγματι, μπορεί κανείς να πει, να πει ότι είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ε, του τώρα ανεψόμενου κλάδου και θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Ακούγοντα την Επιτροπή, πιστεύω ότι η Κομισιό θα πρέπει να προσπαθήσει να είναι ακόμα πιο φιλόδοξη στην προσέγγιση που θα ακολουθήσει εν ώψη των επόμενων διασκέψεων τηλεπικοινωνιών. Γιατί όταν τόσο γρήγορα κινείται η τεχνολογία, αυτή η ITU παγκόσμια διάσκεψη ραδιοπικοινωνιών συνέχεται κάθε τέσσερα χρόνια νομίζω. Αυτό το έχουμε κληρονομήσει από την δεκαετία του 30, του 40, που ήταν διαφορετικά εντελώ τα πράγματα. Ο κόσμο ήταν διαφορετικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευελιξία. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και το θέμα των συχνοτήτων. Πρέπει να έχουμε άνοιγμα στον τομέα αυτό. Οι πολιτικοί πάντοτε χρησιμοποιούν φράσει να λένε ότι το σήμερα ξεκινάει, το αύριο ξεκινάει από σήμερα κτλ. Στον τομέα αυτό όμω αυτό ισχύει κυριολεκτικά. Τώρα θα προετοιμάσουμε τη διάσκεψη του 2015 και έχετε, ε, πρέπει τουλάχιστον να έχετε φιλοδοξίες ώστε να αποκομίσουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο από αυτή την παγκόσμια διάσκεψη. Γιατί εμεί θέλουμε η Ευρώπη να είναι στην πρώτη γραμμή τη παγκόσμια εξέλιξη ό,τι αφορά τι λεπικοινωνίε και τα παγκόσμια σύρματα δίκτυα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν συζητάμε και την κρίση χρέου, αυτό είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση για μα να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ακόμα πιο φιλόδοξη πρέπει να είναι η προσέγγιση και για την ευελιξία, αλλά και για να έχουμε την παγκόσμια ηγεσία στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέκμαρκα. Τώρα εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Κατρίν Τροτμάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπα, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνίων μπορεί να φαίνεται άκρος τεχνικό ε, και στήρο ή στεγνό αν θέλετε, αλλά αν ε, λάβουμε υπόψη μας τη μαζική χρήση των smartphones ε, και την ανάγκη χρήσης περισσότερων συχνοτήτων για τις κινητές επικοινωνίες και πολλές φορές ζητήματα που τα αναλαμβάνουν φορείς διαιτησίας, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι θέματα τεχνικά μόνο, αλλά και εμείς οι νομοθέτες πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους ανάπτυξης αυτών των νέων τεχνολογιών, διατηρώντα ταυτόχρονα τις ήδη φυστάμενες χρήσεις ε, φάσματος, ραδιομετάδοση παραδείγματο χάρη. Πρόκειται για πεπερασμένες ε, ε, δυνατότητες. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη δυνατή χρήση του ραδιοφάσματος για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μελλοντικές εφαρμογές. Και αυτή η παγκόσμια διάσκεψη ραδιοπικοινωνιών του χρόνου που θα καθορίσει και την ατζέντα του 2015 πρέπει πραγματικά να έχει ως αποτέλεσμα μια ευρωπαϊκή ομόφωνη θέση απέναντι ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Πρέπει λοιπόν να τοποθετηθείτε και σε σχέση με τις απόψεις των κρατών μελών, ώστε η Ευρώπη να είναι ένας ε, φορέας που δεν θα μπορεί να παρακάψει κανείς ε, στο παγκόσμιο πεδίο των ραδιοεπικοινωνιών. Δεν είναι θέμα ανταγωνιστικότητας. Μιλάμε για ένα τομέα ικανό να δημιουργήσει θέσεις εργασίας ε, και να προκαλέσει ανάπτυξη. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες πολλές φορές το έχουμε πει αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί ότι ο τομέας αυτός έχει μεγάλο δυναμικό για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη αλλά αγνοείται το δυναμικό αυτό. Θα μπορούσαν όμως να αναπτυχθούν συνέργειες με άλλους τομείς, τον τομέα των μεταφορών, λοιπόν διαστημική πολιτική έρευνα. Αυτή λοιπόν η διάσκεψη που εγγράφεται ε, στη συνέχεια όλων αυτών των συζητήσεων που είχαμε για το διελεκτρικό φάσμα πρέπει να γίνει απογραφή όλων των χρήσεων του φάσματος για να ξέρουμε ακριβώ ε, τις ζώνες που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες. Δεύτερον, το πολύ ακαθόδε ζήτημα των παρεμβολών που πρέπει να λυθεί, χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα, ε, εξωτερικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας ε, δημιουργούν προβλήματα τα οποία πρέπει να υπερπηδήσουμε. Επίση, προσπάθειε για εναρμόνιση και συντονισμένη ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγματι, βλέπουμε να εξελίσσονται οι θέσει των κρατών μελών που και στην αρχή τους προκαλούσε ρίγη και η λέξη απλά εναρμόνιση. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας, κυρία Επίτροπε, ε, για να καταλήξουμε στους στόχους που έχουμε συζητήσει διαμακρών. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τροτμάλη. Ο πρόεδρος εκ μέρους ε, της ομάδας Άλντε τώρα για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Λένα Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σε αυτή την εποχή της κρίσης χρειαζόμαστε όλα τα εργαλεία που έχουμε για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και να γίνει η Ευρώπη ανταγωνιστική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα του φάσματος ε, και οι τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παραδείγματο χάρη για την ψηφία, για το ψηφιακό πρόγραμμα. Πρέπει να αναπτύξουμε την αγορά και να αναπτύξουμε λύσεις ε, τεχνολογίας πληροφορική και επικοινωνιών που θα βοηθήσουν ε, την Ευρώπη να βγει από την κρίση. Ε, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική δημοκρατία, έξυπνες μεταφορές, έξυπνη μέτρηση της ε, ενέργειας, έξυπνα δίκτυα. Πολλά από αυτά είναι δύσκολα και πολλά από αυτά μπορεί να είναι και αδύνατο να επιτευχθούν εάν δεν ε, επιτύχουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις απαραίτητες διεθνείς συμφωνίες όπως είναι οι συμφωνίες της ΕΤΙΓΙΟΥ για το ραδιοφάσμα. Δεύτερον, η Επιτροπή εδώ έχει ένα σημαντικό καθήκον. Πρέπει να διασφαλίσει ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, θα εκπροσωπηθεί σωστά στην διάσκεψη της ITU. Για πρώτη φορά έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπροσωπεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πολιτική του ραδιοφάσματος, παραδείγματος χάρη, που ψηφίσαμε το Μάιο στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι τμήμα της βάσης ε, για, ε, για το ψηφιακό πρόγραμμα και για την Ευρώπη του 2020, για την ανταγωνιστική Ευρώπη με νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Θα συνεχίσουμε να θεσπίζουμε νέους κανόνες σε αυτό το τομέα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ε, τρόπο να επιτευχθεί η συνοχή μεταξύ τη ε, νομοθεσία μα και του διεθνού ρυθμιστικού πλαισίου. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή ε, να διαμορφώσει και να επιδιώξει μια σαφή, μια συνεκτική στρατηγική και να εξασφαλίσει αυτή τη νέα διάσταση στι διαπραγματεύσει αυτέ. Αναμένω από την Επιτροπή ότι θα υπεραμενθεί των αρχών τη διαφάνεια και τη προσωπική ακαιρεότητα, ακριβώ όπω έχουν θεσπιστεί στο πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ την κυρία Εκ. Τώρα η κυρία Λάμπερτς έχει το λόγο εξ ονόματος της, ε, των Πρασίνων. Ah, non, non, ο κύριος Λάμπερτς. Ah, je vous ai pas vu, Δεν σας είχα δει αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στο σημείο που σταμάτησε η Κατρίν Τόρτμαν. Νομίζω ότι το πρώτο στοιχείο για μας ε, είναι το φάσμα, όπως ε, ε, είπες και εσύ Κατρίν πολύ σωστά, είναι ένα δημόσιο αγαθό ε, και επομένως προϋποθέτει ε, καλή συλλογική διαχείριση ε, από, τις, από τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να είναι ή να θεωρεί ότι είναι ιδιοκτήτης του φάσματος. Δεύτερον, αποδεχόμενοι ότι πρόκειται για ένα σπάνιο ε, ε, κοινό αγαθό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο. Πρώτον λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε την ε, παρούσα χρήση του φάσματος. Επομένως να κάνουμε μία, έναν κατάλογο λεπτομερή της χρήσης του φάσματος και βεβαίως από την άλλη πλευρά το να χρησιμοποιείται το φάσμα 2% των δυνατοτήτων του φυσικά δεν θεωρώ ότι είναι μια αποτελεσματική χρήση. Επομένως ένα κατάλογο της παρούσας χρήση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της χρήση αυτής. Τρίτον, Πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό χωρίς σύνορα ε, και εδώ θα ήθελα όπως και ο Γκίναρ να ε, το διασυνδέσω με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αντιμετωπίζομαι εμείς στις χώρες μας Ευρωπαίοι πολίτες βέβαια αλλά ο καθένας προερχόμενος από τη χώρα του αντιμετωπίζομαι έναν εθνικό εγωισμό που λέει ότι αυτό το αγαθό είναι δικό μας, η Ευρώπη δεν έχει να ανακατευτεί καθόλου σε αυτό αλλά ε, θα πρέπει να βρούμε έστω και σε βαθμό επικουρικότητας την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα του φάσματος με ευρωπαϊκό τρόπο ξεπερνώντας τους εθνικούς εγωισμούς. Αυτά ήταν τα τρία σημεία τα οποία ήθελα να θίξω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμπερτ και σας ζητώ συγγνώμη ακόμα μία φορά. 1,5 λεπτό κύριος Βλασάκ παρακαλώ. Από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητών Μεταρρυθμιστών. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nejprve bych chtěl zdůraznit, že považuji za vysoce Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Θέλω να τονίσω ότι θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις διαπραγματεύσει για τα διάφορα σημεία της μείσιας διάταξης τη διάσκεψης αυτής την επόμενη χρονιά. Χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση ε, για τις κινητές τηλεφωνίες και για τις υπηρεσίες ε, στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράμματος και για την πολιτική του ραδιοφάσματος ε, για τα 800 MHz. Ε, χρειάζεται ομοιομορφία και για τη διαχείριση των πτήσεων και για, την, ε, για τις κινητές τεχνολογίες. Θέλουμε να αυξήσουμε την ε, ταχύτητα του δικτύου και να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή τεχνολογιών για την προστασία του συστήματος Galileo και άλλων συστημάτων ραδιοπλοήγησης για την εναέρια κυκλοφορία. Είναι σημαντικά τα έξυπνα συστήματα και οι επιστημονικές δραστηριότητες. για πολλούς τομείς της πολιτικής όπως είναι η αλλαγή του κλίματος. Η χρησιμότητα του ραδιοφάσματος είναι μεγάλη για την κοινωνία και υπάρχει και στρατηγικός και συνολικός παγκόσμιος χαρακτήρας. Τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης θα πρέπει να προωθήσουν την περαιτέρω εξέλιξη, εξέλιξη της τεχνολογίας ευρεία ζώνης Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για ένα λεπτό ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών το Φεβρουάριο του 2012 θα μελετήσει την μεταρρύθμιση των ε, τωρινών ε, κανονισμών και αυτό φυσικά σχετίζεται με τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτείνουν τις δικές τους προτεραιότητες διότι είναι πλήρη μέλη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διάσκεψη ως οντότητα Άρα θα προωθήσει τους στόχους και τις προτεραιότητες της μέσω των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στο σημείο 117 του προγράμματος, δηλαδή χρήση του ραδιοφάσματος ανάμεσα στα 700 και 862 MHz που ε, είναι κατάλληλο δηλαδή για τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Επίσης το σημείο 118 για το σύστημα Galileo, επίσης το σημείο 120 ε, για τα ε, μετεωρολογικά μπαλόνια αερόστατα 25 ε, συγκεκριμένα σημεία στο, στην ημερήσια διάταξη ενδιαφέρον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κέρια σημασία να βρούμε ένα διεύλο επικοινωνία, να έχουμε του κατάλληλου εκπροσώπου στη διάσκεψη που θα επιληφθούν των ζητημάτων και θα πάρουν αποφάσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσει ε, ε, εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Ερχόμαστε στον κατάλογο των αγορητών. Η κυρία Τικάου θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά.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 Ε, κυρία Επίτροπε, στα πλαίσια της παγκόσμιας διάσκεψης ε, ραδιοεπικοινωνιών της ε, ITU θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα πλαίσια του, της, των ραδιοεπικοινωνιών σε όλες τις χώρες μέλη ή μη μέλη. Επομένως, ο, ο ρόλος αυτής της παγκόσμιας διάσκεψης του 2012 είναι πάρα πολύ σημαντικός τα ε, συμβαλόμενα μέρη βεβαίως θα εκφράσουν ε, ε, ενδιαφέρον και το οποίο θα άπτεται συμφερόντων μετρολογικών έρευνας του διαστήματος, βιομηχανίας, οικονομίας κτλ. Το ζήτημα είναι να προωθήσουμε εμείς από τη δική μας πλευρά όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική. Εμείς θα έχουμε 25 στοιχεία τα οποία θα αναφέρονται στο φάσμα, ε, στη χρήση του φάσματος, ε, την εγγύηση ε, του φάσματος, την πλοήγηση, του συστήματος πλοήγησης Γαλιλαίου, τα μετεωρολογικά αερόστατα, την, το, το σύστημα ασφάλειας τα οποία, το οποίο θα έχουν ε, τα ε, πλοία λοιπά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προστατεύσει κυρίως στα πλαίσια του προγράμματος Γαλιλαίο τις, τις παρεμβολές με άλλα συστήματα. Μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των, της αλλαγής από 1504 σε 1505 MHz και επίσης μας ενδιαφέρει ε, όλος ο τομέας της αεροπορίας ε, και ε, είμαστε σε θέση με τον τρόπο αυτό να βελτιώσουμε τις αερομεταφορές. Θα πρέπει πάντως να υπάρξουν και τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά ε, όσον αφορά την χρήση του 1215 ε, ε, και βεβαίως και του GPS του συστήματος Γαλιλαίου. Το πρώτο αφορά τους δορυφόρους που θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τις ερμητοφορές στην Ευρώπη. θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Υποστηρίζω τις θέσεις που ήδη εκφράστηκαν και πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο και στην ηγεσία αυτών τα οποία πρέπει να γίνουν ε, σε αυτό το τομέα. Για να είμαστε ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο ως Ευρώπη θα πρέπει να τονίσουμε τον τομέα των υπηρεσιών και την κοινωνία που θα βασίζεται, την οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση και γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα που αφορούν την δυνατότητά μας σε αυτό το τομέα. Θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ε, στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τροπολογίες της ημερήσης διάταξης αυτής της παγκόσμιας διάσκεψης ε, και θα πρέπει ε, η θέση μας να αντικατοπτρίζεται σε αυτά τα οποία θα προτείνουμε. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά και στρατηγικά τη δύναμή μας. Ακόμη θέλω να τονίσω την αρχή τη επικουρικότητας ω μία από τι πιο σημαντικέ αρχέ που θα μα επιτρέψει ε, να προωθήσουμε τα συμφέροντα των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, σπάνια συμβαίνει αυτό. όσοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, θα τον πάρουν Προς το παρόν έχει ζητήσει ο κύριος Κάστλερ το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα για το θέμα αυτό να υπενθυμίσω και στην Επιτροπή και σε όλους εμάς στην Ευρώπη πόσο σημαντικό είναι για μας το τομέα των τεχνολογιών ε, της ε, ε, ραδιοεπικοινωνία, ε, να βρισκόμαστε στην κορυφή των εξελίξεων και να είμαστε μία από τι μεγάλε δυνάμει σε ολόκληρο τον κόσμο, να είμαστε υπερήφανοι για την τεχνογνωσία μα, διότι έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε ε, θέματα όπω τον Γαλιλαίο. Υπάρχουν πολλά σημεία, πολλοί τόποι στους οποίους προάγεται η εργασία του Γκαλιλαίου και στη δική μου την περιοχή στην Νιρεμβέργη και έχουμε τεράστιο δυναμικό και τεχνογνωσίας και χρειαζόμαστε υποστήριξη για να συνεχιστεί αυτή η έρευνα ούτως ώστε αυτά τα προγράμματα στο μέλλον να εδραιώσουν και να αναπτύξουν τη θέση μας παγκοσμίω. Γι' αυτό τονίζω την παράκλησή μου να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε αυτά τα μεγάλα συστήματα όπως ε, τον Γαλιλαίο και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε την ε, ηγετική θέση και την ανεξαρτησία μας ε, παγκοσμίω. Και στην επόμενη διάσκεψη των ραδιοεπικοινωνιών αυτό θα πρέπει να τονιστεί επαρκώς από όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ήθελα να ρωτήσω άλλοι συνάδελφοι, άλλες συνάδελφες θέλουν να πάρουν το λόγο πρωτού τον δώσω στην Επίτροπο και κλείσει η συζήτηση. Οπότε, ε, Miss Commissioner, you have the floor. Ευχαριστώ. Ε, σημειώνονται ραγδαίε εξελίξει σε αυτό το τομέα. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό και όλα είναι συναρπαστικά. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ε, θα υπάρξει φυσικά ε, σημείο τη μερίσια διάταξη για την πολιτική ραδιοφάσματο, για την κατάσταση ανά τον κόσμο. Εξετάζουμε το θέμα του ραδιοφάσματο για τι ευρυζωνικέ κινητέ συνδέσει και πάνω από 1000 MHz θα έχουν εναρμονιστεί, το οποίο είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Η Επιτροπή δεν μπορεί το 2012 να εκπροσωπηθεί στη διάσκεψη. Και γι' αυτό επιζητούμε συζήτηση με, με τα κράτη-μέλη για τη μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος. Ε, φυσικά θα επιδιώξουμε δια το μέγιστο δυνατό συντονισμό στην Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε και τον απολογισμό ε, και πρόκειται για μια πρόταση που εντάσσεται στην πολιτική ραδιοφάσματο ε, τη Ευρώπη. Ε, φυσικά, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου για την εκπόνηση τη στρατηγική ε, ραδιοφάσματο, διότι έχει μια στρατηγική διάσταση. Ε, το θέμα των δικτύων ε, και όλα τα συναφή ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, ανακοίνωσή μας που συζητούμε, συζητείτε εδώ σήμερα και θα συζητήσετε και στο μέλλον φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το σημείο για μας και άρα προσβλέπουμε με ανυπομονησία σε μελλοντικέ συζητήσεις και συνεργασία για το θέμα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για το θέμα της συζήτησης αυτής ε, από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Έληξε εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι, λίγο αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα για ένα διάλειμμα μέχρι τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ.